Η Επιτροπή ΕΝΒ έχει διαβιβάσει την εξή διόρθωση σε ένα κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του κανονισμού, αυτή η διόρθωση θεωρείται εγκεκριμένη εκτός αν εντός 24 ώρων από την ανακοίνωσή της μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές ζητήσουν να ψηφιστεί, να τεθεί μάλλον σε ψηφοφορία. Η διόρθωση υπάρχει στην ε, σελίδα, ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος της θα δημοσιευθεί στα, επόμενα, στα πρακτικά της επόμενης συνόδου.